και θα στηρίξουμε επίση και την πολιτική και οικονομική ανάπτυξη τη χώρα. Σα ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε. Μισάρια. Σα ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Επίτροπε. Θα ψηφίσουμε, αφού πλέον έλξει η συζήτηση, θα ψηφίσουμε ε, μόλι ολοκληρωθεί η συζήτηση για τα κατεπήγοντα. Και περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο τη ημερησιά διάταξη, που είναι η συζήτηση για το Γουαντάναμο, απεργίε πείνα των κρατουμένων. Όπω γνωρίζετε, θα έχουμε κάποιες παρεμβάσει, αλλά μπορεί να υπάρξει μια διπλή ερμηνεία εδώ. Δηλαδή, ίσως κάποιοι σκεφτούν ότι είχαμε συζήτηση χωρίς ψηφοφορία. Έτσι είχα καταλάβει εγώ πάντως ε, ότι τώρα θα συζητούσαμε και τη, σε κάποια άλλη μεταγενέστερη ε, σύνοδο θα ψηφίζαμε. Ήταν και μια πρόταση από τον συνάδελφο Σβόποντα, ε, την οποία με υπόψη της η διάσκεψη των Προέδρων και που καταρτίζει την σχέδια Δεν ξέρω αν θα ψηφίσουμε στην επόμενη ε, σύνοδο που για μένα είναι το φυσιολογικό, ή κάποια άλλη στιγμή. Τώρα δεν κατάλαβα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αποφασιστεί. Εμεί είπαμε θα συζητήσουμε για το Γκουαντάναμο, αλλά θυμάμαι ή κατάλαβα ότι πρόκειται για συζήτηση χωρί ψήφισμα. Νομίζω ότι πρέπει να γραφεί στα πρακτικά αυτό, για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση. Δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουμε καθόλου δεν θα ψηφίσουμε τώρα. Έχει αναβληθεί η ψηφοφορία. Έχει ξαναγίνει αυτό και με άλλε συζητήσει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο σε μια σειρά από συναδέλφου που είναι οι συντάκτε των ψηφισμάτων. Ο φίλο Ροή Ταβάρη είναι ο πρώτο. Έχετε 1,5 λεπτό για την παρέμβασή σα, κύριε Ταβάρη. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητή κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα κι εγώ, ξεκινώντα, όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, ότι φυσικά και πρέπει να ψηφίσουμε για το Γκαντάναμο και λυπούμε πολύ που δεν θα ψηφίσουμε σήμερα, γιατί πάνω από 150 άτομα βρίσκονται σε αυτό το στρατόπεδο χωρίς να έχουν καταδικαστεί εδώ και χρόνια, ε, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, δεν έχουν δικαστεί αυτά τα άτομα και δεν μπορούν να έχουν και την ε, υπηρεσίε τη υπεράσπιση. Πολλοί λοιπόν βρίσκονται σε απεργία πείνα, κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους ε, καταναγκαστικά τρέφονται ορισμένοι εξ αυτών και πραγματικά η κατάσταση είναι κατεπίγουσα. Είναι επονίδιστο. Είναι επονίδιστο το ότι αποφασίσαμε να έχουμε μόνο συζήτηση και όχι ψήφισμα, διότι το Κοινοβούλιο είναι ένας χώρος συζήτησης και ο στόχος είναι να περάσουμε κάποια μηνύματα. Δεν ήρθαμε εδώ για να πιούμε τον καφεδάκι μας, θέλουμε να δείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι έχουμε ένα μήνυμα να δώσουμε. Θέλουμε λοιπόν ψήφισμα και με το ψήφισμα αυτό θα ζητήσουμε από τις Ηνωμένε Πολιτείες, διότι Ξέρουμε ότι στην σύλληψη και παράνομη κράτηση ε, των φλεξιμένων συνεισέφεραν και συνεργάστηκαν γι' αυτό και κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξουν εξέλιξει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Και ολοκληρώνοντα, εκφράζω την λύπη μου για το γεγονό ότι ορισμένοι συνάδελφοι εκμεταλλεύτηκαν ε, την ε, βομβιστική επίθεση στην Βοστόνη, η Μαλιλέγγυο με τα θύματα, για να ζητήσουν αναβολή τη ψηφοφορία αυτού του ψηφίσματο. Δεν θα πρέπει ποτέ τέτοιου είδου συμβάντα να τα χρησιμοποιούμε ω μέσα πολιτική πολιτική πίεση για να επιτύχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Πρέντα, ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εμείς λυπούμεθα γιατί η συζήτηση έπρεπε να αναβληθεί. και θα πρέπει να κρατήσουμε ενό λεπτού σιγή για τα θύματα της Βοστόνης. Ευχαριστώ κύριε Πέρα. Τη διευκρίνηση αυτή έπρεπε να την θέσετε στην αρχή της συνεδρίασής μας το πρωί. Φυσικά και είμαστε αλληλέγγυοι με τα θύματα αυτού του ατυχήματος. Έχει το λόγο για 1,5 λεπτό η κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι την στιγμή που θάβει η Αμερική τα θύματα της φαγής της Βοστόνης δεν μπορούμε με επιπολαιότητα να αναφερθούμε στο Γκουαντάναμο αλλά πρέπει να αναφερθούμε. Εδώ και 11 χρόνια οι φυλακισμένοι στη φυλακή αυτή βιώνουν συνθήκες που γνωρίζουμε, συνθήκες εκτός δικαίου Θυμάμαι ότι ο κύριος Έλμαρ Μπρόκ μετά από μια επίσκεψη στην Κουαντάνα μου είπε είδα τι σημαίνει έλλειψη δικαίου. Θα σας θυμίσω επίσης κάτι το τρομερό για μένα, την δίκη του Άντερς Μπρέιβικ, ο δολοφόνος αυτός, ο οποίος προχώρησε στη σφαγή του Όσλο τον Ιανουάριο του 12. Θα θυμάστε την αυστηρότητα, τη λιτότητα, την αξιοπρέπεια της δίκης αυτής και αυτή την τρομερή ε, στάση των δύο εισαγγελέων οι οποίοι πήγαν και έδωσαν το χέρι τους στον ένοχο. Γιατί έπρεπε να αντιμετωπιστεί ο ένοχος αυτός όπως οποιοδήποτε άλλος ε, υποψήφιος ένεχος. Σε αυτήν την απόλυτη δεοντολογία, σε αυτή την εσωτερική δύναμη του δικαίου βρίσκεται και ο τρόπος αντιμετώπισης, ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης ε, της τρομοκρατίας με την αξιοπρέπεια και ε, το δίκαιο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρξει νόμος στο, ε, στο Γκουαντάναμο όλοι είναι ε, αθώοι έως ότου καταδικαστούν. Αν σεβαστούμε την αξιοπρέπειά τους τότε ε, φοβάμαι ότι η τρομοκρατία θα μας υπερνικήσει. Φυσικά οι Αμερικανοί δεν έπρεπε να πάθουν αυτό το οποίο έπαθαν και στο μαραθώνιο της Βοστόνης να θυμίσω όμως ότι στο Γκουαντάναμο ο Ομπάμα επιτέλους πρέπει να σεβαστεί τις υποσχέσεις του και δεν του το επιτρέπει το Κογκρέσο και η Ευρώπη θα πρέπει να μπορέσει κάποιους από αυτούς τους κρατουμένους να τους υποδεχθεί στα εδάφη της. Γιατί δεν τους κατηγορούν για τίποτα, πολύ απλά. Έχει ζητήσει ο Χάνς Πέτερ Μάρτιν να σας κάνει μια ερώτηση. Θέλετε να απαντήσετε. Έχετε το λόγο κύριε Μάρτιν, 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, συμφωνώ μαζί σας. Πιστεύω πως πρέπει να είμαστε συνεπείς. Όμως τώρα όπως μιλήσατε για την Ορβηγία, ε, μου θυμήσατε τι έγινε το 1972 Στου Ολυμπιακού αγωνέ του Μονάχου και είπαμε «The games must go on». Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Συζητούμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν πρέπει λοιπόν να παραμελήσουμε καμία λεπτομέρεια. Πρέπει να το συζητήσουμε διεξοδικά. Euh, Ευχαριστώ τον Χάνς Πέτερ Μάρτιν για την ερώτησή του. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να υπάρξει μια συμβιβαστική λύση. Η συμβιβαστική λύση είναι ο καλύτερος τρόπος και έτσι εργαζόμαστε και εμείς στο Κοινοβούλιο. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε. Δεν το επιθυμούσαν οι συνάδελφοι και γι' αυτό πρότεινα αυτή την συμβιβαστική λύση ή ψηφοφορία να γίνει αργότερα. Έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε όλοι τι πρέπει να γίνει σε σχέση με το Γουαντάναμο. Ευχαριστώ. Έχει το λόγο η κυρία Σάκε. Για ένα λεπτό το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Όπως και οι Ηνωμένε Πολιτείες και εμείς γνωρίζουμε τι σημαίνει η τρομοκρατία και την καταπολεμούμε. Προσπαθούμε να υπερασπιστούμε επίσης και τις κοινωνίες μας από επιθέσεις από το εξωτερικό, αλλά θα πρέπει να απαγορεύσουμε να υπάρχουν διαβρώσεις από το εσωτερικό. Δεν μπορεί να παίρνουν όλα τα μέτρα χωρίς συνέπειες. Η Αμερική ε, είναι ε, σύμμαχός μας, πολύτιμος, αλλά δυστυχώς παραβιάζει βασικές αρχές του δικαίου ε, όπως η προϋπόθεση φυσικά της αθωότητας και άλλες βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι αξίες διακρίνουν τις ανοιχτές κοινωνίες από τις περιορισμένες κοινωνίες. Ο νόμος ο Αμερικανικός για την αντιμετώπιση της δημοκρατίας δυστυχώς είναι κάτι το πάρα πολύ αρνητικό. Αν αυτά τα οποία έκαναν οι Αμερικανοί τα έκαναν οι Αγίπτοι, οι Ηνωμένε Πολιτείε πρώτες θα τα καταδίκαζαν. Και ταυτόχρονα ε, το ότι δεν μπορούν οι δικηγόροι να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην επικοινωνία με τους πολίτες τους, με τους πελάτες τους, συγγνώμη, είναι απαράδεκτα πράγματα. Πρέπει η φυλακή αυτή να κλείσει αμέσως. Οι δημοκράτες θα πρέπει να στοχεύουν στα υψηλότερα επίπεδα. Ο Στόλτεμπεργκ, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, μετά τη σφαγή του Μπράιβικ είπε ότι η βία δεν αντιμετωπίζεται παρά με τη δημοκρατία. Ευχαριστώ συνάδελφε. ενάμιση λεπτό για την κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Σόνι και εκνευρίστηκα λίγο περισσότερο. Είναι στο χαρακτήρα μου. Την Τρίτη δημοσιεύθηκε μια έκθεση στις Ηνωμένε Πολιτείες καταδικαστική για τα συστηματικά βασανιστήρια στον Κουαντάναμο. Πράγματι παρά τις υποσχέσεις που είχε δώσει ο Ομπάμα το 2008 λόγω της αρνητικής τάσης του Κογκρέσου, η βάση του Γκουαντάναμο είναι πάντα εκεί και η κατάσταση των ανθρώπων που είναι εγκλειστοί εκεί είναι ανησυχητική. 130 φυλακισμένοι αυτή τη στιγμή κάνουν απεργία πείνας, αντιμετωπίζονται με απαράδεκτο τρόπο, τους στερούν το πόσιμο νερό, τους τρέφουν με βία και την προηγούμενη Παρασκευή υπήρξε ε, διαφορετικό επίπεδο άσκησης βίας από πλευράς των κρατουμένων Μέχρι τώρα έχουν περάσει από τον Κουαντάναμο 770, 770 περίπου κρατούμενοι. Ε, οι περισσότεροι δεν έχουν κατηγορηθεί. 600 ε, τόσοι είναι ακόμα εκεί, πάνω από 11 χρόνια. 80 ε, από αυτούς θα έπρεπε να είναι ελεύθεροι αλλά δεν μπορούν να φύγουν γιατί δεν έχουν χώρα να πάνε και πράγματι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γίνονται τα πράγματα αυτά έτσι όπως γίνονται και συμφωνώ με την κυρία Ντεκεζέρ. Η βάση του Γκουαντάναμο πρέπει να κλείσει, είναι μελανό σημείο για τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου όπως θέλει να αυτοπροσδορίζεται. Θα πρέπει να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι αυτοί εφόσον δεν έχουν κατηγορηθεί για κάτι. Θα πρέπει να βοηθηθούν για να βρεθεί μια χώρα υποδοχής για αυτούς και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει το ρόλο της και να υποδεχθεί ένα τμήμα αυτών των κρατουμένων. Ευχαριστώ κυρία Βερζιά. Παρακολουθήσαμε ε, αυτά που είπατε προς τον κύριο Σόνικ που είναι ε, δημοκράτης και ευγενέστατος κυρίως και δέχτηκε πραγματικά θετικά αυτά που είπατε. Εξ ονόματος Σοσιαλιστικής Ομάδας ο κύριος Χάουιτ για ένα λεπτό. Είναι τρομερή η τραγωδία που συνέβη στην Βοστόνη αλλά και στο Τέξας. Ναι, λυπούμαστε πάρα πολύ για τα θύματα, όμως πρέπει να συζητήσουμε και να συνεχίσουμε να συζητούμε, γιατί όταν υποφέρει ένας υποφέρουν όλοι. Συνεχίζεται η απεργία πείνας και για ορισμένους οι συνέπειες είναι μη αναστρέψιμες στον Γκουαντάναμο και κάθε μέρα που περνάει κάνοντας απεργία πείνας έρχονται πιο κοντά στο θάνατο. Στις 6 Φεβρουαρίου άρχισαν οι απεργίες πείνας και πιστεύω πως απολύτως σωστά το Κοινοβούλιο σήμερα πρέπει να συνεχίσει αυτή τη συζήτηση. Λαμβάνουμε πληροφορίες ότι 13 από τους απεργούς πείνας ε, ταΐζονται με το ζόρι μέσω σωλήνα και μέσω καθετήρα και πραγματικά είναι καθήκον αυτού του Κοινοβουλίου να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες και να αναρωτηθεί εάν αυτή η μεταχείριση είναι η σωστή. Πρέπει να γίνουν συζητήσεις με το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτικών για να βελτιωθούν οι, κατάστα... για να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης. αυτή η κατάσταση είναι κάτι το οποίο καταδικάζουμε. Arvoisa puhemies. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η τρομοκρατική επίθεση στη Βοστόνη ήταν τρομακτική, όλοι την καταδικάζουμε. Η υπεράσπιση μιας δημοκρατικής κοινωνίας προϋποθέτει να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην περίπτωση του Γκαντάναμο, οι Ηνωμένε Πολιτείε παραβιάζουν σαφέστατα τα ανθρώπινα δικαιώματα με αυτές τις συνθήκες κράτησης. Οι Ηνωμένε πολιτείες ενεργούν απολύτως αντίθετα στις δικές τους αξίες όταν κρατούνται άνθρωποι χωρίς κατηγορία και χωρίς δίκη. 26 κρατούμενοι πρόκειται να απελευθερωθούν όμως αυτό δεν θα γίνει, δεν θα απελευθερωθούν περισσότεροι επειδή δεν υπάρχει άλλος χώρος. Μιλήσατε για δίκαιη δίκη και καλές συνθήκες κράτησης. Η κατάσταση στον, ε, στον Κουαντάναμο είναι μία από τις μεγαλύτερες ντροπέ της παγκόσμιας κοινότητας από την ίδρυσή του έως σήμερα. Ελπίζω πολύ σύντομα οι Ηνωμένε Πολιτείε να αποφασίσουν να κλείσει τον Κουαντάναμο. Ελπίζω να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις Ηνωμένε Πολιτείε στο σκοπό αυτό και ελπίζω αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέτρεψαν στις επικράτειές τους ε, μυστικές φυλακές για ε, κρατουμένους των ΗΠΑ και αυτό το βρίσκω πραγματικά επονίδιστο. Στην ε, μάχη κατά της τρομοκρατίας έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα τα οποία αντιτίθενται στις αξίες τις οποίες η δυτική κοινωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείες υπερασπίζονται και έχουν δεσμευτεί να τηρήσουν. Έχουν γίνει λάθη και αυτά τα λάθη όμως δεν πρέπει να επαναληφθούν. Un minuto para su intervención el señor Schlitter que habla en nombre de los Verdes. Ευχαριστώ πολύ. Όταν ήμουν μικρός μεγάλωσα στις Ηνωμένε Πολιτείε, όπου ήταν όπως ξέρετε η χώρα των ελευθέρων. Έλαβε χώρα πόλεμος του Βιετνάμ. Η παγκόσμια κοινότητα ζήτησε από τις Ηνωμένε Πολιτείες να αποσυρθεί από αυτόν τον πόλεμο. Όμως ε, τότε υπερασπίστηκαν και αξίες όπως το κράτος δικαίου και ισότητα. Υπήρξαν άνθρωποι που υπερασπίζονταν τις Ηνωμένε Πολιτείες. Τώρα ε, λαμβάνει χώρα πόλεμος κατά της τρομοκρατίας και τώρα παρατηρούμε βασανιστήρια, επιθέσεις, παράνομες κρατήσεις, όλα αυτά να γίνονται μυστικά και κλεισμένων των θυρών. Έχει έρθει η ώρα να βοηθήσουμε τον Αμερικανικό λαό να υπερασπιστεί τη δημοκρασία και να σεβαστεί το κράτος δικαίου παρά να συνεχίσει τον πόλεμο της ε, τρομοκρατίας και αντί για χώρα των ε, ελευθέρων να, το, να λέμε χώρα των φυλακισμένων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να εδράζονται και ο σεβασμός τους σε πανανθρώπινες αξίες. Φυσικά καταδικάζονται φαινόμενα όπως η παράνομη φυλάκιση και αυτό θα πρέπει να ισχύσει και για τους κρατούμενους του Γκουαντάναμο είναι γεγονός ότι άνω των ε, μισών αυτών που βρίσκονται εγκλειστοί εκεί είναι γνωστό ότι είναι αθώοι και όμως παρόλα αυτά εξακολουθούν να κρατούνται. Αυτό δείχνει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι σε θέση να αποφασίσουν τι θα κάνουν με αυτούς. Το 2009 ο πρόεδρος Ομπάμα είπε ότι θα έκλεινε την φυλακή του Γκουαντάναμο και μάλιστα υπέγραψε ε, δυστυχώς αργότερα την συνέχιση λειτουργίας του στρατοπέδου αυτού συγκέντρωσης ουσιαστικά. Η απεργία πείνας των κρατουμένων μας υπενθυμίζει ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια πολιτισμένη, μια νομικά αποδεκτή λύση στον Κουαντάναμο. Σας ευχαριστώ. εξ των μη γραμμένο του κ. Βάντερ Στουπ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ δυσκολεύομαι κύριε Πρόεδρε να μιλήσω για την κατάσταση στο Guantanamo Bay όταν ε, σήμερα έχουμε την ε, κηδεία των θυμάτων της Βοστόνης. Παρ' όλα αυτά είναι επίκαιρο το ζήτημα. Ε, στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λοιπόν Έχουμε συμπεριλάβει το σημείο αυτό στην μια διάταξη. Γνωρίζουμε ότι στον Καντάνα, Μουμπέ υπάρχουν κρατούμενοι οι οποίοι υποφέρουν. Δεν έχουν γίνει σεβαστά πολλά, πολλές, δεν έχουν γίνει πολλές από τις αρχές ε, του διεθνούς δικαίου και σίγουρα υπάρχουν και κατάφορη παραβίαση πολλών ε, διατάξεων της διεθνούς δικαίου όπως το habeas corpus. Έχουν ε, ξεκινήσει λοιπόν κάποιες πολύ άσχημες διαδικασίες η απεργή πείνας δεν είναι κάτι το οποίο με αφορά πάρα πολύ γιατί είναι ένας προ... τρόπος ε, προσέγγισης προσοχής και βλέπουμε ότι είναι και επιτυχημένος. Θα μπορούσα να πει ότι είναι ένα αμερικανικό πρόβλημα, εσωτερικό και ότι δεν θα έπρεπε εμείς να βάλουμε στη σφικοφολιά το χέρι μας. Δεν θα πρέπει, ε, πιστεύω, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λειτουργεί ως χώρο ε, υποδοχής ε, πρώην κρατουμένων του Γκαντάνων. Πολλοί νέοι μουσουλμάνοι στις χώρες μας θα τους δουν ως μάρτυρες του ανθρώπου αυτού και ε, ως ένα λόγο για να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Φυσικά και τα άτομα αυτά θα πρέπει να απελευθερωθούν σε περίπτωση που δεν έχουν κατηγορηθεί για τίποτε. Και η Αφρικανική Ένωση και ο ΑΣΕ επίση θα πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρο, πάμε τώρα στου ε, υπόλοιπου ομιλητέ, που δεν είναι παρά ένα, ο κύριο Ρέπο. Ένα λεπτό έχετε, κύριε Ρέπο. Κύριε Πρόεδρε, το σαλαπτό του Καντάνα μου είναι να αγκάθι στο πλευρό του πρόεδρου Ομπάμα και ένα πάρα πολύ σοφερό παράδειγμα των ε, υπερβολών ε, της, ε, διεθνούς, του Διεθνούς Αγώνα κατά της Τρομοκρατίας. Ο πρόεδρος Ομπάμα υποσχέθηκε να το κλείσει το Γκουαντάνο το 2009. Είναι ακατανόητο το γεγονός ότι κρατούνται εκεί για 11 χρόνια άνθρωποι χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία ή να έχουν δικαστεί. Αυτό αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Δυστυχώς, οι αρχές ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φαίνεται να μην εφαρμόζονται στην εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Στο διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ΗΠΑ θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως θέμα συζήτηση, πιστεύω, και τον Κουαντάναμο. Οι απεργοί πείνα ε, ουσιαστικά ε, ζητούν βοήθεια. Ε, η κίνησή τους είναι μια κραυγή βοήθεια. Δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν και θα πρέπει και η θέση κοινότητα του Σταυρού να έχει πρόσβαση. Ευχαριστώ, λέει ο Έχουμε τέσσερις συναδέλφους στη διαδικασία Catch Παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομη, να μην περιέσουμε το ένα λεπτό καθένα για να τηρήσουμε το ωράριο που έχουμε. Λοιπόν, πρώτος, ο κύριο Μασίπ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ στηρίζω τα λόγια που άκουσα εδώ από το φίλο μου, το Ρουί Ταβάρης από τη Βερονίκ Ντεκάιζερ, από το Ρέπο, τον Χάουιτ, φυσικά, διότι είναι σοβαρότατο αυτό το οποίο γίνεται στον Κουαντάναμο και ποτέ δεν πρέπει ε, να το ξεχνάμε εμείς οι δημοκράτες ε, του κόσμου. Ναι, όμως είναι κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, είναι ίσως το πιο σοβαρό, η πιο σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να θυμόμαστε ότι, ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ε, αυτές ε, που ε, δεν επιτρέπουν στην Κούβα να συνεχίσει. Κι είναι μόνο έδαφος που δεν μπορεί να πατήσει η Αμερικανική μπότα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν πρέπει να φύγει από το Γιβραλτάρ, δεν πρέπει να φύγει η Τουρκία από τη Βόρεια Κύπρο, δεν πρέπει το Μαρόκο να φύγει από τη Δυτική Σαχάρα. Διότι ο πολιτισμός μας, κύριε Μασίπ, δυστυχώς Τελείωσε ο χρόνος σας. Ο κύριος Γότσον, ο επόμενος ομιλητής. Για 12 χρόνια οι πρακτικές ανάκρισης παραβιάσεις ε, στις συνδίκες κράτης του Καντάναμου ουσιαστικά αντιτίθενται ε, στο δικαίωμα για την επιδίωξη ευτυχίας και της ζωής. Μόνο τρεις από τους κρατούμενους έχουν καταδικαστεί. Το ίμιση έχουν αθωωθεί ε, και ζουν λέει ο Ντικ Τσένεϊ, πάρα πολύ καλά, τρέφονται, έχουν ό,τι θέλουν ε, στη διάθεσή τους. Αυτό αποτελεί πραγματικά προσβολή στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είναι ένα γκούλαγκ ε, της σύγχρονης εποχής και έχει υποσχεθεί ο Ομπάμα θα το κλείσει. Ε, τέσσερα χρόνια μετά όμως ε, σε μια πράξη απόγνωσης ε, βλέπουμε τους κρατούμενους να κάνουν απεργία πείνας. Εμείς είμαστε υπέρ της ηθικής ακαιρεότητας. Σίγουρα είμαστε στο πλευρά των Αμερικανών για την ε, καταπολέμηση της δημοκρατίας και θρυνούμε τα θύματα της Βοστόνης, αλλά θα πρέπει η αδικία αυτή να ξέρουν ότι τελικά δεν θα αποτρέψει τους εχθρούς ε, της ελευθερίας, αλλά θα στρατολογήσει και άλλους. Ευχαριστούμε κύριε Γουότσον. Ο κύριος Ρωμέβα τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω 43 άτομα, όπως λένε οι επίσημοι, ή 130 με βάση της Οργάνωσης των Δικαιωμάτων, ε, πρέπει να τύχουν του σεβασμού μας. Ε, θα πρέπει να έχουμε μία ε, γνωμοδότηση για αυτούς. Κάποιοι πραγματικά δίκαια είναι σε απεργία πείνας και παραλαμβάνω ότι όλες οι χώρες πρέπει να τηρούν τη διεθνή νομοθεσία. Και αυτό σίγουρα έχει να κάνει και με τη ΣΥΠΑ. Και είπα, τη ΣΥΠΑ ισχύει. Το 9, ο ε, πρόεδρος Ομπάμα που πήρε βραβείο Νόμπελ όπως ε, πέρυσι η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι θα το κλείσει. Ε, τα προεδρικά όμως δικαιώματα και τα προνόμια δεν τα χρησιμοποίησε για να σταματήσει κράτηση αυτών των 160 κρατουμένων πολέμου. Σίγουρα δεν μπορούμε, όπως είπε και ένας άλλος από το ΕΛΚ, να εκμεταλλευόμαστε και να χρησιμοποιούμε τη, τα θλιβερά και ε, τραγικά συμβάντα της Βοστόνης για να ξεχάσουμε αυτή την περίπτωση του Γκουαντάναμου. Ε, ευχαριστώ, πρόεδρος. Τώρα θα κλείσει η κυρία Γκέριγκερ Ντε Έντεμπεργκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το 2009 και το 2013 επίσημα είπε η Αμερικανική κυβέρνηση ότι θα κλείσει την βάση του Ογκαντάναμο. Δυστυχώς δεν το έχει κάνει. Υπάρχουν σε αυτή τη φάση 160 κρατούμενοι ε, οι οποίοι είναι ύποπτοι για συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες. Για τους περισσότερους από αυτούς καμία κατηγορία δεν απαγγέλθηκε και καμία δίκη δεν έγινε. Το προηγούμενο Φλεβάρι η μισοί από αυτούς τους φυλακισμένους ξεκίνησαν μια απεργία πείνας. Υπήρξαν και συγκρούσεις ανάμεσα στους δεσμοφύλακες και τους φυλακισμένους. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση δείχνει ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πρέπει αμέσως να περάσουμε στο κλείσιμο του Γκουαντάναμο και να μεταφερθούν όλοι οι κρατούμενοι στις χώρες προέλευσης. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα πρέπει να κλείσουμε λοιπόν την συζήτηση με την παρέμβαση της Επιτρόπου της κυρίας Μέλστρομ. Αγαπητά μέλη, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στις φρικτές ε, επιθέσεις στη Βοστόνη και να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών και τις αρχές της χώρας αυτής. Η απεργία πείνας ξεκίνησε πριν δύο μήνες, την προηγούμενη εβδομάδα, είπαν οι Αμερικανικές αρχές ότι 43 από τους 160 αρνήθηκαν να τραφούν. Τώρα οι αριθμοί ακριβώς είναι θέμα συζήτησης, αλλά πάνω κάτω έχει η κατάσταση έτσι. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχει μια απελπισμένη θα έλεγα ακατάσταση, γιατί πολλοί από αυτούς παραμένουν φυλακισμένοι χωρίς κατηγορίες και χωρίς δίκες. 11 ε, από αυτούς έχουν χάσει τόσο μεγάλο βάρος που έπρεπε να τραφούν ε, καταναγκαστικά. Αυτό είναι ένα θέμα που θέτει προβλήματα και ε, ηθικά και νομικά. Υπάρχει το δικαίωμα φυσικά του ασθενούς, υπάρχουν τα δικαιώματα του να δεχθεί ή να μην δεχθεί τροφή, αλλά η καταναγκαστική διατροφή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναλύεται από τις δικαστικές αρχές κατά περίπτωση. Πάντως παρακολουθούμε το θέμα αυτό με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όπως ακριβώς είπε και ο Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ερυθρού Σταυρού. Οι συνθήκες λοιπόν αυτές και η ένταση που επικρατεί στην ε, μονάδα αυτή μας ανησυχεί. Είμαι πεπισμένη ότι η καλύτερη και πιο ανθρώπινη κατάσταση είναι να ξεκινήσει η πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει στο πλήρες κλείσιμο της μονάδας κράτησης στον Κουαντάναμο. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι η βάση θα έλεγα της πολιτικής μας παρέμβασης εναντίον της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εναντίον της αφαίρετης κράτησης και το Συμβούλιο και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν εκφράσει τις απόψεις τους γύρω από αυτό ζητώντας να κλείσει τον Κουαντάναμο και θα το επαναλάβουμε αυτό σήμερα λέγοντας ότι η βασική ευθύνη είναι στις Ενωμένε Πολιτείες. Εμείς ανταποκριθήκαμε σαν φίλος, σαν εταίρος στο αίτημα για σύνδρομη από πλευρά της Αμερικανικής κυβέρνησης Ήδη από το 2009 συζητήσαμε το κοινό πλαίσιο και γι' αυτό δεχθήκαμε 20 τέος κρατουμένους στην περιοχή αυτή, στην βάση αυτή. Από τότε το Αμερικανικό Κογκρέσο στα πλαίσια του νόμου του 2012 και του 2013 παρατείνουν την κράτηση χωρίς δίκη και έτσι περιορίζουν την δυνατότητα της ε, κυβέρνησης να μεταφέρει ε, τους κρατουμένους του Γκουαντάναμο. Επανειλημμένα και σε υπουργικό επίπεδο εμείς έχουμε συμμεριστεί με τους Αμερικανούς τις ανησυχίες μας για τη συμβατότητα των προβλέψεων αυτών με την διεθνή τάξη, τον διεθνή νόμο και τις αρχές της διατλαντικής συνεργασίας. Είμαστε οι στενότεροι σύμμαχοι και φίλοι των Ηνωμένων Πολιτειών Πρέπει να τους βοηθήσουμε για να καταπολεμήσουμε όλοι μαζί την τρομοκρατία, αλλά να υποστηρίξουμε επίσης και τις προσπάθειες της Αμερικανικής κυβέρνησης για να κλείσει επιτέλους η φυλακή του Γκουαντάναμο. Ευχαριστώ Επίτροπε με την δική σας παρέμβαση. Κλείνει η συζήτηση αυτή και θα περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Έχουμε